der präsident! επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα έγγραφα τα οποία έχουν εγκριθεί είναι στη διάθεσή σας. Έχετε αντιρρήσεις. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε λάβει μια αίτηση του ΕΛΚ για την αντικατάσταση της κυρίας Σουίτσα.